σαν επικοδομητικό τόσε πολλέ φορέ. Επομένω, πείστε την κυρία Τιμοσέγκο να κάνει αυτά που έκανε και ο κύριο Γιανακόβη. Ευχαριστώ, κύριε Σφόμποντα. Ακολουθεί ο κύριο Μιγκάσκι για ένα μισή λεπτό. Ε, κύριε Πρόεδρε, Επίτροπε,